Morning everybody and please be seated. Please be seated in silence. Παρακαλώ καθίστε και κάντε και λίγο ησυχία. Να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Didier Reinders, υποψήφιο επίτροπο, τον οποίον καλώς ορίζουμε θερμά. Καλώς ήρθατε αγαπητέ. Η ακρόαση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο επιτροπές μας, καθώς ε, το χαρτοφυλάκιο της δικαιοσύνης είναι αρμοδιότητας ε, και των δύο επιτροπών μας. όπως έχει ε, καταρτιστεί σύμφωνα με την επιστολή της ανάθεσης της κυρίας Φόντερ είναι σαφές ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δύο επιτροπών μας λοιπόν. Πρώτα απ' όλα το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει στόχο να διασφαλίσει το κράτος δικαίου ε, εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης και της του προτινόμενου διευρυμένου μηχανισμού κράτους δικαίου που επηρεάζει την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ε, αυτά περιγράφονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, που ετέσαν ισχύ μαζί με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας πριν από 10 χρόνια και είναι δεσμευτικό δίκαιο σύμφωνα με την ομολογία του ΔΕΚ. Επίσης, επηρεάζει τον αντίκτυπο που έχει η χάρτα αυτή στην ιδιωτικότητα, στην ψηφιακή εποχή, που είναι επίσης ένα από τα χαρτοφυλάκια που έχει σχεδιάσει η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην Μελλοντική Επιτροπή επίσης. Επηρεάζει και το πακέτο εφαρμογής ε, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και το σημαντικότερο, βεβαίως, πρέπει να φροντίσουμε εμείς να ε, βελτιωθεί η κατάσταση της δικαστικής ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αμοιβαία αναγνώριση. για να μπορέσει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ε, που έχει εννέα τον αριθμό. Οπότε θα πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. που θα λειτουργήσει από το 2020. Έτσι θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ε, νόμοθεσίας, έτσι ώστε το εταιρικό δίκαιο να προωθεί μια στρατηγική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, αποτελεσματική συνεργασία επίσης στους τομείς ε, αστικού και ποινικού δικαίου έγκαιρη και σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε, να σας υπενθυμίσω ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό παίζει ρόλο κεντρικό στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε για να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, όπως είναι η πολιτική βούληση και η νομική εντολή που έχουμε στον τίτλο 5 της συνθήκης που βασίζεται όπως σας είπα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη την αμοιβαία αναγνώριση και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πάλι ποτέ κριτήρια της Κοπενχάγης ε, που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε τότε το δίλημα της Κοπενχάγης ε, περί δεσμευτικών ε, αρχών και αξιών που θα είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη και ε, ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι ισχύει του εθνικού και δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Δίνουμε τώρα τον λόγο στην συμπρόεδρο την κυρία Λούση Νέτσιγκα πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Thank you very much. Um, it's, it's a delight to be here. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Ρέντερς. Ελπίζω να είναι επικοδομητική συνάντηση για όλους μας. Ε, η Επιτροπή Γιούρη πολύ ε, χαίρεται που είναι παρούσα στην ε, συνεδρίαση αυτή και θα επικεντρωθούμε σε θέματα προστασίας του καταναλωτή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια διαδικαστικά θέματα τη σημερινή συνεδρίαση. σύμφωνα με το παράρτημα 17 του κανονισμού, που περιέχει τις ε, κατευθυντήριες γραμμέ για έγκριση τη ε, για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα εξετάσει το Κοινοβούλιο την ανεξαρτησία και την καταλληλότητά τους, καθώς και τις γνώσεις τους στα σχετικά χαρτοφυλάκια. Το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει ερωτηματολόγιο στον ε, Οριστέντα Επίτροπο ε, με κάποιες εισαγωγικές γενικές ερωτήσεις και κάποιες πιο συγκεκριμένες. Ο ε, Επίτροπος έχει απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και έχει διανεμηθεί, έχουν διανεμηθεί απαντήσεις σε όλους τους βουλευτές και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Επίσης δεν υπήρξε αντίρρηση όσον αφορά την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η συζήτηση θα διεξαχθεί ω εξή Ο οριστή επίτροπος ε, θα κάνει μια εισαγωγική ε, παρουσίαση 15 λεπτών και μετά από αυτό θα ακούσουμε 25 ερωτήσεις από του ευρωβουλευτέ. Η συζήτηση αυτή θα γίνει ως εξής. 5 ε, λεπτά στον καθένα, 1 λεπτό ερώτηση, 2 λεπτά απάντηση και κατόπιν δεύτερη ερώτηση 1 λεπτό με 1 λεπτό για την απάντηση επίσης. Οι πρώτες 7 ερωτήσεις ε, θα τεθούν από τους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων, ε, ενώ ο επόμενος γύρος 18 ερωτήσεων θα γίνει από τους υπόλοιπους σύμφωνα με το μέγεθος των πολιτικών ομάδων και μία ερώτηση για ανεξάρτητο βουλευτή. Και στο τέλος θα έχουμε 5 λεπτά για την τελική απάντηση του ε, ορίστε επιτρόπου. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας, αλλιώς δεν θα υπάρχει χρόνος ε, να τεθούν ερωτήσεις και να απαντηθούν σωστά. Ε, σας προειδοποιώ λοιπόν ότι αν ξεπεράσετε το χρόνο σας θα αναγκαστώ να σας διακόψω και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. ερμηνεία παρέχεται σε 23 γλώσσες.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 Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα το πρωί ενώπιον σα και μάλιστα χαίρομαι ακόμη περισσότερο διότι βλέπω πολλά οικία πρόσωπα σήμερα. Θα ήθελα να σα μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούμε από κοινού εφόσον ε, με εμπιστευτείτε στο πλαίσιο τη αποστολή ε, την οποία μου ανέθεσε η οριστήσα ε, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Φοντερ Συγκεκριμένα μου ανέθεσε να διευθύνω το έργο τη Κομισιόν σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, τη δικαιοσύνη και την προστασία των καταναλωτών. Όπω γνωρίζετε, Έχω διατελέσει ευρωβουλευτή, μάλλον ε, βουλευτή και σέβομαι ιδιαίτερο στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι θεωρώ ότι έχετε σημαντική συνεισφορά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε την παρέμβασή μου, με δύο πιο προσωπικά ε, σχόλια. Το πρώτο ε, είναι κάτι που μην ιδιαίτερο προσφυλέσει η θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Πριν από 20 χρόνια για πρώτη φορά ε, ανέλαβα καθήκοντα υπουργού. Τότε η Ευρώπη ήταν διαιρεμένη και αγωνιζόταν για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της πτώσης του τείχου. Στα τελευταία 20 χρόνια άλλαξαν πολλά πράγματα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και ευτυχείς με τα όσα έχουν επιτελεστεί και πραγματοθεί εδώ στην Ευρώπη. Διότι έχουμε πολιτικές, νομοθεσία για την ευημερία των πολιτών. Δεν ε, ε μου ένα στον άλλο για εδάφη. Διατηρούμε την πολυμορφία μας μέσω του πολιτισμού, των γλωσσών μας. Αν λοιπόν επιβεβαιωθώ ως Ευρωπαίος Επίτροπος, ε, δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ μαζί σας με αποφασιστικότητα για την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είμαι από αυτούς που θέλουν περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αν θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή σε μια παγκόσμια τάξη που εξελίσσεται, θα το πετύχουμε μόνο αν είμαστε ενωμένοι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε είναι πως ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι όλο και πιο κατακαιρματισμένος και ασταθής. Οι αξίες μας απειλούνται από όσους θέλουν να επανέλθουν σε εθνικιστική, λαϊκιστική ρητορική, κάτι που θα έπρεπε να ανοίξει στο παρελθόν. Οι αξίες μας απειλούνται από κράτη τα οποία θέλουν να κυριαρχούν και όχι να συνεργάζονται. Βασικό μας χρέος και καθήκον είναι να προστατεύσουμε τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία. Όμως και να προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες, ε, τη στήριξή μας ε, στα πολυμερή όργανα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην κοινωνική πρόοδο. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι για να προασπίσουμε παντού το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό απαιτεί να πράξουμε το αυτό και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και το δεύτερο σχόλιο είναι ακόμη πιο προσωπικό. Στις 14 Σεπτεμβρίου, το προηγούμενο Σάββατο, έμαθα ότι εδώ και μήνες ε, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο εσκεμένα προσπαθεί να με αποσταθεροποιήσει και να με βλάψει. Έχει καταφέρει σοβαρές καταγγελίες ε, σε βάρος μου και δημοσία έχει δηλώσει ότι θέλει να με εμποδίσει να γίνω Ευρωπαίος Επίτροπος. Έχω αρνηθεί όλους τους ισχυρισμού του ε, που ανέφερε ο τύπος ε, και ο δικηγόρος με έλαβε, είχε επαφές με την εισαγγελία για να λάβει γνώση του δικογράφου. 27 Σεπτεμβρίου ο Βασιλικός Εισαγγελέας, συμφωνώντας πλήρως και με τον Γενικό Εισαγγελέα, εισαγγελέα έβαλε στο αρχείο ε, αυτό το δικόγραφο και δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια επειδή δεν υπήρξε κανένα, καμία αξιόπινη πράξη. Το ίδιο κάνει ο δικηγόρος μου ε, και στη νέα ε, προσφυγή που έκανε το συγκεκριμένο άτομο. Δυστυχώς κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι μπορεί να πέσουμε θύμα μια τέτοιας κακόβουλης επίθεσης. Δεν θα ευχόμουν σε κανέναν να ζήσει αυτά τα οποία οι συγγενείς μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, η σύζυγός μου και εγώ προσωπικά ζούμε τις τελευταίες αυτές 15 ημέρες. Το κράτος δικαίου είναι μεταξύ άλλων το τεκμήριο της αθωότητας. Και γι' αυτό ήθελα να σας τα πω αυτά τα πράγματα για να είμαι ξεκάθρο απέναντί σα. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, ακριβώ 20 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 1999, πρώτο επίτροπο αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων ανέλαβε ο Αντώνιο Βιτορίνο. Θα ήθελα να το αποτίσω φόρο τιμή, όπω και στου διαδόχου του και ιδίω στην Βέρα Γιούροβα και τον Φραν Τίμερμαν, για το σθένο του, για την αποφασιστικότητά του. Αν γίνω επίτροπο, θα συνεργαστώ πολύ στενά μαζί του. Χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που η κυρία Φοντρελάιν με πρότεινε ε, για να αναλάβω τα θέματα δικαιοσύνης αλλά και προστασίας καταναλωτών και σεβασμού κράτους δικαίου. Τρεις πτυχές του χαρτοφυλακίου μου που είναι στενά συνδεμένες μεταξύ τους. Το χαρτοφυλάκιο εδράζεται στις αρχές της εμπιστοσύνη, της ένταξη, της ισότητα. Ε, Αυτό είναι ο γνώμονα για καθεμία από αυτέ τι τρει πολιτικέ. Θα είναι ε, στον πυρήνα. Κυρίε ε, και κύριοι βουλευτέ, αυτό ισχύει ιδιαίτερω για το κράτο δικαίου. Θεωρώ ότι πρέπει να προβάλλουμε τι αξίε μα ε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και να τι τηρούμε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω Επίτροπο Δικαιοσύνη θα συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο για τι αξίε και τη διαφάνεια, έτσι ώστε το κράτο δικαίου να τηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα συνεργαστώ στενά με την Επίτροπο Αρμόδια για την Γειτονία και την Διεύρυνση για να διασφαλίσω την συνοχή Τη προσέγγιση αυτή στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερος αγαπητό. Ως υπουργό των Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχω ζητήσει για μια πιο έχω ζητήσει μια πιο ενεργή δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει και να προστατεύσει το κράτο δικαίου. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία και σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα χωρί σεβασμό για το κράτο δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αποτελεσματικά μόνο αν προστατεύονται από ανεξάρτητα δικαστήρια. Η δημοκρατία προστατεύεται μόνο εάν τα δικαστήρια μπορούν να διασφαλίσουν την ελευθερία τη έκφραση τον πλουραλισμό των ΜΜΕ και του κανόνε των εκλογών. Το κράτο δικαίου δημιουργεί αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τόσο σημαντική για την εσωτερική αγορά μας. Πιο σημαντικό ακόμα, έχει μεγάλη σημασία για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η ευθύνη μας είναι να διαφυλάξουμε το κράτος δικαίου σε κάθε κράτος μέλος. Έχουν παρουσιαστεί αρκετές ιδέες, μεταξύ των οποίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας δοθούν τα εργαλεία για να εμβαθύνουμε στο έργο αυτό. Τον Ιούλιο η Κομισιόν παρουσίασε τις προτάσεις της για έναν συνολικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κράτους Δικαίου. Θα προωθήσει μια κουλτούρα κράτους δικαίου, θα προλάβει την εμφάνιση ανησυχιών και θα ανταποκρίνεται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Θα προωθήσω αυτό το έργο και του χρόνου θα ξεκινήσουμε με μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ετήσια και προληπτική. Έτσι θα έχουμε μια ετήσια έκθεση και τον πίνακα βαθμολογίας δικαιοσύνης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Η παρακολούθηση θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά θα εμβαθύνει περισσότερο στα κράτη-μέλη εκείνα στα οποία έχουν αναγνωριστεί ιδιαίτερη κίνδυνη. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδώσω στην διασφάλιση της αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης αυτής της παρακολούθησης και το πώς θα οικοδομηθεί διάλογος και θα έχουμε βέλτιστες πρακτικές για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Έχει σημασία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εμπλέκονται πλήρως. Πρέπει επίσης να συντονιστούμε καλύτερα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε τους ίδιους στόχους και ιδεώδη. Πιστέψτε με, δεν θα διστάσω να δράσω όποτε κινδυνεύει το κράτος δικαίου. Δεν θα συμβιβαστώ όταν διακυβεύεται η δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προσαρμογή των δικαστικών συστημάτων στην ε, Γρήγορε αυτέ αυτές εξελίξει είναι μία, μείζον προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία. Είναι σημαντική η ενίσχυση τη δικαστική ε, συνεργασία σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Το δικαίωμα να ζει κανεί, να εργάζεται κανεί στην Ένωση με πλήρη σεβασμό τη ελευθερία τη διακίνηση θα πρέπει να διατηρηθούν. Επίση πρέπει να διαφυλάξουμε την πολυμορφία μα ε, εγγυόμενη ταυτόχρονα ότι οι διαφορετικέ νομικέ παραδόσει δεν θα συνιστούν εμπόδιο στην ελευθερία στην ασφάλειά μα. Δεσμεύομαι ότι θα κάνω πάντο δυνατό ώστε να ενισχύσω το κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων. Αξιότιμοι βουλευτέ, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, θα συνεχίσω να παρακολουθώ την εφαρμογή του και να συνεργάζομαι στενά μαζί σα και με τα κράτη-μέλη, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το μηχανισμό αυτό. Πρέπει να δούμε προσεκτικά τι χρειάζεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση τη εξολόγηση τη συμμόρφωση που είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε κατά πόσο απαιτούνται διαδικασίε και με βάση την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα δω επίσης κατά πόσο να χρειάζεται να καταθέσω πρόταση για αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης. Επίσης ε, θα ήθελα να δω πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν ε, και οι συνθήκες στα σοφρονιστικά ιδρύματα στην Ένωση και θα διερευνήσω την ιδέα να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την προσωρινή κράτηση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μία άμεση ε, δουλειά που έχω να κάνω είναι να καταστεί επιχειρησιακή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θέλω να χαιρετήσω το ρόλο που διαδραματίσατε ε, για να υπάρξει συμφωνία σε ό,τι αφορά το, ε, τη νέα επικεφαλής. Ήρθα σε επαφή πρόσφατα με την κυρία και είμαι πεπισμένος ότι θα φέρει σε πέρα στην αποστολή της. Επίσης, ε, πρέπει να σωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες για να εξυγχρονίσουμε τα νομικά δικαστικά συστήματα, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα είναι πιο αποτελεσματική η δικαιοσύνη, πιο προσβάσιμη στους πολίτες. Πρέπει όμως να φροντίσουμε η εφαρμογή του δικαίου και ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Πρέπει να είναι και μπορεί να είναι η περήφανη που είναι παγκόσμιο ηγέτη σε θέματα προστασία δεδομένων και σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρώπη. Η προτεραιότητά μα λοιπόν είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα να πήχουν πλήρους προστασία στην ψηφιακή εποχή. Θα εργαστώ μαζί σας για να βρούμε τη χρυσή τομή. Θα φροντίσουμε να υπάρξει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε και να προωθήσουμε επίσης τα πρότυπα και τις αξίες μας σε διεθνές επίπεδο. Θα εργαστώ επίσης με τους συναδέλφους για να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες και ηθικές επιπτώσεις τη τεχνητής νοημοσύνη. Χαίρομαι που μας δίνει δυνατότητες η νέα τεχνολογία, αλλά θα πρέπει προτεραιότητά μας επίσης να είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, η εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη ε, είναι η βάση για την προστασία του καταναλωτή ε, στη δική μου προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο και εκτός. Θέλουμε βιωσιμότητα στην κοινωνία και σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς και τα επιχειρηματικά και καταναλωτικά μοντέλα. Το επιχειρηματικό δίκαιο μπορεί να ε, βοηθήσει την ε, οικονομία και θα πρέπει οι καταναλωτές να κάνουν σωστές επιλογές. Οι καταναλωτές από μόνοι τους, ο καθένας ξεχωριστά, δεν έχει ε, πολύ δύναμη, αλλά μαζί είναι πολύ ισχυροί αν μπορούν να ενεργούν ε, σε εμπεριστατωμένη βάση και αυτή η αγοραστική δύναμη μπορεί να δημιουργήσει μια βιώσιμη οικονομία. Γι' αυτό ακριβώς θα ασκήσω πίεση για γρήγορη υιοθέτηση της πρότασης για τις ε, συλλογικές για τις ε, συλλογικές ε, προσφυγές. οι δυνατότητες αυτές είναι απαραίτητες για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα πρέπει να εφαγρυπνούμε όσον αφορά τα προϊόντα ε, διότι θα πρέπει ε, να έχουμε την ίδια ενιαία ποιότητα όλων των προϊόντων, ώστε να μην παραπλονείται ο καταναλωτής. Και σημείο αφετηρίας ε, είναι να έχουμε ασφαλή προϊόντα, είτε αυτά παράγονται στην Ευρώπη είτε αλλού. Θα εξετάσω την αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Επίσης θέλω σαφείς κανόνες ε, για την ευθύνη των ε, προμηθευτών ε, στα προϊόντα που πολλούνται επιγραμμικά. Τέλος, σκοπεύω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου. Μεγάλο, μεγάλος όγκος καταναλωτικού δικαίου έχει οθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να φροντίσουμε τώρα ε, να εφαρμόζεται σωστά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, σε σχέση με τους διεθνείς εταίρους μας. Κύριε Συμπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, μίλησα για το τι έχουμε πετύχει ε, νωρίτερα τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε περήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει. Έχουμε όμως και υποχρέωση προς το μέλλον. Αυτό ξεκινά με το να είμαστε ε, έτοιμοι να ακούμε και εγώ θα σας ακούω σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Υπάρχουν εκατομμύρια νέοι που κατεβαίνουν στους δρόμους ζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι πηγή έμπνευσης για μας και μας καλούν να αναλάβουμε δράση από κοινού έχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να πετύχουμε. Ελπίζω να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Κύριε Οριστέντα, Επίτροπε Ρέιντερς. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Ε, θα ακούσουμε ε, συνολικά 25 και θα έχουμε την ε, ίδια δομή. Δύο λεπτά ε, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά πρώτη απάντηση, ένα λεπτό αντίδραση από τον Ευρωβουλευτή και άλλο ένα λεπτό από τον ε, Οριστέντα Επίτροπο. Θα ξεκινήσουμε ως συνήθως από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πέντε λεπτά λοιπόν έχει ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ και τον κύριο Ανδρέη Χαλίκη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Ρεντέρς, για, την, για τον ορισμό σας και να ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική ερώτηση, συγκεκριμένα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ε, με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών κανόνων. Κανόνων που άπτονται του κράτους δικαίου, που εσείς ο ίδιος είπατε ότι είναι ακρογωνιαίος λήθος. Στοιχείο το οποίο ευνοεί την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Και στοιχείο που αφορά όλους τους τομείς της δικαιοσύνης καθώς και της αστυνομικής συνεργασίας και των οικονομικών πολιτικών που με την εσωτερική αγορά. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού στην πράξη και τι βήματα ε, σκέφτεστε να κάνετε για να εξασφαλίσετε το σεβασμό του κράτους δικαίου όταν, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, υπάρχουν κράτη τα οποία θέτουν από αμφισβήτηση τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Βλέπουμε παραδείγματα παρενόχλησης ε, και κατάχρησης ε, ε, απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς. Βλέπουμε ότι και η ελευθεροτυπία ή η ελευθερία λόγου απειλούνται. Πώς μπορούμε λοιπόν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταχρήσεις. Να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να τηρείτε το χρόνο σας, διότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι να τηρούμε το χρόνο ομιλίας. Ένα λεπτό για αρχική ερώτηση, δύο λεπτά για απάντηση και μετά άλλο ένα λεπτό για να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλίτσικ για την ερώτησή του. Ο οργανισμός για το κράτος δικαίου θα είναι σίγουρα στο επίκεντρο της εντολής μου. Όπως γνωρίζετε, εδώ και πάνω από τρία χρόνια στο επίπεδο του Συμβουλίου ζητώ να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αξιολόγησης από μοντήμου στο peer review και ξέρετε τον Οκτώβριο του 2006 υπήρξε και ένα έγγραφο για την επιτήρηση του κράτους και ε, η έκθεση του Ιουλίου σίγουρα η ανακοίνωση αυτή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα διευθύνω λοιπόν ε, τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα περιοριστούμε όμως το κράτος δικαίου. Μιλάμε για τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ, για τη δημοκρατία ε, και θέλω ε, ετησίως να κάνω τον απολογισμό. Θα καταθέσω και τον πρώτο χρόνο στη, στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο ε, την έκθεση αυτή. Υπάρχει αυτή η εργαλειοθήκη, αλλά υπάρχουν και άλλα. Ε, υπάρχει το άρθρο 7, παραδείγματο χάρη, το οποίο ε, ενεργοποιήθηκε ε, για την Πολωνία από την Κομισιόν και η Ουγγαρία εξε, αντιμετώπισε την κρίση σας και υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε βέβαια να έχουμε ένα διάλογο με τις ε, χώρες αυτές. Θα το πράξω και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβώ ε, στις χώρες αυτές όταν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω. Έχουμε τον Γκρέκο, έχουμε την Επιτροπή της Βενετίας και άλλα εργαλεία για την προσαρμογή της νομοθεσίας ε, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καλύτερα. Δηλαδή ο μηχανισμό αυτό είναι μόνο ένα εργαλείο. Υπάρχουν και πολλά άλλα σε την εργαλειοθήκη που έχει στη διάθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μην χρειάζεται να ξανακινήσουμε τα δικασία του άρθρου 7. Θα το δούμε όμως αυτό συν το χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Ρέιντερς. Ε, κύριε Χαλίκη, άλλο ένα λεπτό έχετε για να αντιδράσετε σε αυτό που ακούσατε. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τα ξεχωριστά αυτά μέσα που αναφέρατε. Είναι σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών κτλ. Όταν υπάρχει κάποια απειλή όμως ε, θα πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε άμεσα. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα μέσα. Ε, άλλο ένα λεπτό κύριε Ρέιντερς. Ναι, είπα ότι υπάρχουν ε, διαδικασίε επί στο πλαίσιο τη εργαλειοθήκη. Σίγουρα υπάρχει όμω ένα διάλογο πολύ σημαντικό, ο οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί όπω και εγώ ζητούμε να υπάρχει ε, σύνδεση, να υπάρχει μια, μια σχέση ε, μεταξύ χρηματοδότης κράτους δικαίου, ε, μια αιρεσιμότητα. Και ελπίζουμε οι συνομοθέτες να καταλήξουν συμφωνία από αυτό, διότι αυτό θα μας δώσει πράγματι τη δυνατότητα να μπορούμε να αναλάβουμε άμεσα δημοσιονομική δράση να αναστείλουμε κάποια δημοσιονομικά μέσα ή και να τα καταργήσουμε ενδεχομένω ε, όταν ένα κράτος γενικευμένα ε, δεν τηρεί τις δεσμεύσεις τους και τις υποχρεώσεις τους ό,τι αφορά το κράτος ε, δικαίου. ίσως βέβαια αυτό να μην είναι τόσο αμυγός για τη δικαιοσύνη συζήτηση και να αφορά πιο πολύ τα δημοσιονομικά, αλλά σίγουρα αυτό που ζητάτε θα το πράξουμε. όταν υπάρχουν παραλήψεις σίγουρα θα δράσουμε αναλόγως. Προχωράμε τώρα ε, στον κύριο Τιέμο Βόλκεν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρέιντερς, ε, καλώς ήρθατε ε, στην ακρόαση αυτή. Λυπάμαι που δεν αναφέρατε την ε, ε, επιχειρηματική βιωσιμότητα και τη δέουσα επιμέλεια. Για μας η διαφάνεια είναι στοιχείο κλειδί ε, για την επιχειρηματική λογοδοσία όσον αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή έχουμε οδηγία για την υποβολή οικονομικών εκθέσεων, ε, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται μεγάλες επιχειρήσεις ε, να υποβάλουν ε, στοιχεία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως αναθεώρηση για να είναι κατάλληλη για, το για να πετύχει το στόχο της. Σκοπεύετε να τροποποιήσετε την οδηγία αυτή, να θυμάστε ότι σήμερα πάνω από 84 ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα S&D και εγώ προσωπικά συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από απλά κατευθυντήρες γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά έχετε, κύριε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ανέφερα στην εισαγωγή μου την υποχρέωσή μας να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό. Όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, είμαστε προσιλωμένοι στην επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, σε επίπεδο ΟΗΕ και εσείς μιλήσατε για συγκεκριμένους ε, κανονισμούς. Υπάρχουν ε, κάποιες μη οικονομικές ε, πληροφορίες που πρέπει να υποβάλουν ε, οι, οι συγμένες επιχειρήσεις, αλλά πράγματι στο επιχειρηματικό δίκαιο είναι ίσως σημαντικό να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα, να έχουμε άλλες απαιτήσεις. Εάν θέλουμε μια πραγματικά βιώσιμη πολιτική, θα πρέπει να ζητήσουμε από όλε τις επιχειρήσεις να σκεφτούν τον τρόπο που σκέφτονται το κοινωνικό συμφέρον. Το κοινωνικό συμφέρον δεν είναι μόνο ένα βραχυπρόθεσμο όραμα, είναι και μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αφορά το κλίμα, αφορά τις τοπικές κοινότητες, το περιβάλλον, ε, άλλες ομάδες ενδιαφερομένων ε, πέρα από τους μετόχους. Είμαι πολύ προσιλωμένος στη συνεργασία μαζί σας ε, και με το Συμβούλιο για να εισάγουμε νέε απαιτήσει ε, στο επιχειρηματικό δίκαιο. Εσείς μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν ε, και άλλα. Ε, υπάρχουν κάποιες απαιτήσει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά είμαι βέβαιος ότι πρέπει να τροποποιήσουμε σημαντικά, ουσιαστικά, το επιχειρηματικό δίκαιο, να ζητάμε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική δράση των επιχειρήσεων. Και δεν αρκεί απλά να κατονομάζουμε. Εάν μια επιχείρηση πρέπει να εξηγήσει, να παρουσιάσει ένα πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα, θα πρέπει <clears throat> να ζητήσουμε από την επιχείρηση αυτή πιο αναλυτικές παρατηρήσεις. Ε, Κύριε Βέλκεν, άλλο ένα λεπτό έχετε. Ε, κύριε Ρέιντερ, αποφύγατε να δώσετε συγκεκριμένη ερώτηση. Τι συγκεκριμένα βήματα θα αναλάβετε για να φροντίσετε ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, <clears throat> να να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύουν το περιβάλλον. Και τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την πρόσβαση σε νομικά μέσα σε όσους έχουν ζημιωθεί από επιχειρήσεις ευρωπαϊκές και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα σήμερα να δεσμευτείτε σε ένα πλαίσιο που να δίνει σαφή δικαιώματα ε, στους Ευρωπαίους πολίτες και που να διασφαλίζει την εφαρμογή ε, διεθνών συνθήκων, πρότυπα του ΟΣΑ για παράδειγμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου δώσετε σαφή απάντηση στην ερώτηση αυτή. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Η απάντησή μου είναι σαφής. Ναι, φυσικά είμαι προσιλωμένος στους στόχους αυτούς, ε, αλλά σε διάφορα πλαίσια. Τώρα μίλησα για το επιχειρηματικό δίκαιο. Άκουσα τις παρατηρήσεις σας ε, για την δυνατότητα αντίδραση από πλευρά των πολιτών. Ε, όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Είμαι διατεθειμένος όμως να εργαστώ πάνω στην καλύτερη νομική βάση ώστε να φροντίσουμε όλοι οι οικονομικοί παράγοντες να Ε, τηρούν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και είμαι βέβαιος ότι αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορες νομοθετικές πράξεις. Είμαι απόλυτα προσιλωμένος σε αυτό και η απάντησή μου ήταν ε, σαφής. Με ρωτήσατε θα κάνω κάτι και είπα ναι. Προχωράμε στο... Περνάμε στον κύριο Μίχαλ Σιμέκα, εκπρόσωπο τη Ρινιού. Έχετε ένα λεπτό για την ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας υποψήφια επίτροπε. Λοιπόν, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και η δημοκρατία είναι όλα βασικά σημεία για την επιβίωση των πλουραλιστικών κοινωνιών μα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα όμω είναι κάποιε κυβερνήσει στα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν την πλειοψηφία του για να υπονομεύσουν τον πλουραλισμό και να εδραιώσουν την εξουσία τους μέσω του νόμου. Οπότε το θέμα είναι ευρύτερο, όπως το αναγνωρίσατε και εσείς. Ως Επίτροπος λοιπόν αρμόδιος για αυτόν τον συνολικό μηχανισμό θα επεκτείνεται τον τίτλο του για να καλύπτει το πλήρες πεδίο του άρθρου 2, δηλαδή δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι, συμφωνείτε ότι βασικό λόγο για τον οποίο αργεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι διαφορετικέ προσεγγίσεις των θεσμικών οργάνων, πολλέ προτάσει, πολλέ ιδέε, πολλά μέτρα θα σκεφτείτε έναν ενιαίο μηχανισμό που θα περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα και θα λάβει μορφή δεσμευτικής διοργανικής ε, συμφωνίας με βάση αυτά τα οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο το 2016. Κύριε Ρεντέρ, έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση αυτή για τον μηχανισμό και το ποιο θα είναι ο ιδιώτη τρόπος να έχουμε μια συνολική προσέγγιση όχι μόνο για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ακριβώς συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Μίλησα για την πλουραλισμό και τον ΜΜΕ. Αλλά θα γνωρίζετε ότι η Κομισιόν επίσης σκοπεύει να συντάξει μια έκθεση για την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα συνεργαστούμε Προ μια νέα στρατηγική για την έκθεση για τη δημοκρατία. Θα εργαστώ λοιπόν για το θέμα του κράτου δικαίου, γιατί όπω ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη διαδικασία για να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Το συζητάμε εδώ και κάποια χρόνια εδώ, αλλά και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν για το πώ θα οργανωθεί μια τέτοια διαδικασία. Αλλά είμαι σίγουρο ότι πρέπει να συνεργαστούμε και για να συνεργαστούμε θα πρέπει να οργανώσουμε μία συζήτηση για όλα τα διαφορετικά στοιχεία δηλαδή την έκθεση για το κράτος δικαίου, την έκθεση για την χάρτα και πιθανώς την έκθεση για τη δημοκρατία. Και αυτό ε, σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μια διοργανική συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα είναι επίσημη γιατί ίσως θα καθυστερήσει, αλλά να ξεκινήσουμε αμέσως. Και γιατί όχι, θα προτείνω να οργανωθεί μια ομάδα εργασίας με τα τρία θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο συζητούσε ε, μία έκθεση από μοτίμους, η Κομισιόν επίσης ε, και το Κοινοβούλιο με το κείμενό σας ε, του Οκτωβρίου του 2016 για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την διαδικασία. Βεβαίως θα δούμε πρώτα, πρώτα την έκθεση αυτή, αλλά είναι εύκολο να δούμε την διαδικασία αυτή, όπως είπα, συνολικά, όπως είπατε, δηλαδή κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στην ομάδα εργασία αυτή τους να τον Ευχαριστώ. Κύριε Σημαντικά έχετε άλλο ένα λεπτό για να αντιδράσετε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις και για το ότι δεσμεύεστε να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση και τα όσα υποσχέθηκε η κυρία Φοντελάιεν έτσι ώστε η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο να έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, σύμφωνα με το άρθρο 225. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ρητός ότι αυτό θα ισχύσει και σε αυτό το ζήτημα και στην έκθεση που συνέταξε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2016. Ρωτάω γιατί στη νέα πρόταση της ε, Κομισιόν και στις γραπτές σας απαντήσεις απορρίψατε την ιδέα που πρότεινε το Κοινοβούλιο για ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης ή πάνελ ειδικών που θα αξιολογεί το κράτος δικαίου. Αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν συχνά χρησιμοποιεί ανεξάρτητους ε, ειδικού ακριβώς για την επιβολή των διαφόρων ε, πολιτικών της, διατηρώντας την συνολική πολιτική ευθύνη, οπότε δεν βλέπω κάποιο νομικό ή πρακτικό εμπόδιο για να χρησιμοποιηθούν και εδώ πέρα ανεξάρτητοι ειδικοί. Συμφωνείτε λοιπόν πως ε, έχει κέρια σημασία η εξέταση από ανεξάρτητους ειδικού για να είναι αντικειμενική και ουδέτερη. Σας ευχαριστώ κύριε Ρεντέρς. Έχετε τον λόγο. Δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστούμε με ανεξάρτητους ειδικού. Το κάνουμε. Έχουμε την Επιτροπή της Βενετίας, το Γκρέκο και άλλες ομάδες ειδικών. Αλλά υπάρχει μια ευθύνη της ε, Κομισιόν ενώπιον του Κοινοβουλίου. Οπότε αν έχετε κατά νου και άλλους ανεξάρτητους ε, φορείς ε, που θα μπορούσαμε να συμβουλευτούμε για τέτοια ζητήματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δούμε αν θα φτιαχτεί ένας νέος ανεξάρτητος φορέας με ευθύνη και ίσως ε, χωρίς την ίδια προσέγγιση. Αν είναι να δώσουμε σε ανεξάρτητο φορέα την πλήρη ευθύνη να εκφράζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως περίεργο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Κομισιόν, να έρχεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο να αποφασίζει. Και τελευταία παρατήρηση, βεβαίως αν έχουμε πραγματικό πρόβλημα, υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, έτσι, το δικαστήριο. Και εκεί πέρα ε, αλλάζει υπόθεση. Οπότε δεν άρνουμε ε, την δυνατότητα να συζητήσουμε με ανεξάρτητους ειδικού ε, και ανεξάρτητους φορείς, αλλά όχι να ε, δημιουργήσουμε ένα νέο φορέα. Σας ευχαριστώ κύριε Ρεντέρς. Τώρα είναι η σειρά των πρασίνων. Η κυρία και Μπρικμό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνάπτει πολλές ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της δικαιοσύνης, του εμπορίου, και είπατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξάγουμε τα πρότυπά μας στους διεθνούς εταίρους, ότι θα επενδύσετε και στην εσωτερική και στην εξωτερική διάσταση, ότι θέλετε να βελτιώσετε τη δικαστική συνεργασία και επίσης ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όσων εμπλέκονται σε ποινικέ διαδικασίες και σε ό,τι αφορά την προσωρινή κράτηση. Τώρα, ε, το ερώτημά μου είναι εάν δεσμεύεστε να ε, κάνετε συστηματικά μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πώς ε, θα εξασφαλίσετε την προστασία των δικαιωμάτων αυτών στο πλαίσιο συμφωνιών ε, με την, μεταξύ Europol και των κρατών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αυγής και πώς θα συνεργαστείτε με τους επιτρόπους ε, για τις εμπορικές συμφωνίες και τη μετανάστευση. Κύριε Ρέιντερς, να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι είναι η απάντηση για το κατά πόσον θέλω να γίνουν μελέτε αντικτύπου. Ναι, συμφωνώ, πρέπει να γίνουν μελέτε αντικτύπου για μια σειρά νέων πρωτοβουλειών που αναλαμβάνουμε σε επίπεδο ένωση. Φυσικά και θα πρέπει όταν δεσμευτούμε και έχουμε συζητήσει ε, με εταίρου τρίτα κράτη επίσης ε, να σέβομαστε αυτές τις δεσμεύσεις. θα ήθελα να μπορώ να ενημερώνω το Κοινοβούλιο όπως και το Συμβούλιο σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων. Μελέτη αντικτύπου λοιπόν θα ενταχθεί σε αυτή την ανάλυση. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια θα το κάνω σε όλους τους τομείς, σίγουρα θα το κάνω στους τομείς που άπτονται άμεσα του χαρτοφυλακίου δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να γίνει κοινή δουλειά, όπως είναι προφανές και ε, με άλλους επιτρόπους, ε, δηλαδή στον τομέα των στερικών. Είπατε ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Ευρω Europol και κάποιες χώρες. Πρέπει να προσέξουμε εκεί πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο πλαίσιο της σύναψης αυτών των συμφωνιών. Υπάρχουν και υπηρεσίες ε, που πάγονται στη δικαιοσύνη και με αυτές θα συνεργάζομαι. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να εντείνουμε την, τον προβληματισμό μα ε, για την συμπερίληψη ρητρών των ε, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμπορικέ συμφωνίε. Και αυτό βέβαια αφορά όλε τι πολιτικέ ε, απέναντι στι τρίτε χώρε. Όπω ξέρετε, δεν έχουμε πάντα την ίδια προσέγγιση με όλου του εταίρου μα στο κοινοβούλιο σα.